Σα καλωσορίζω λοιπόν στην κίνη μας συνεδρίαση με την ΤΕΒΕ. Καλωσορίζω την συνάδελφο την κυρία Λίντα Μακάβαν. Λίντα Μακάβαν. Λοιπόν, στην έκθεση για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και το τι μπορεί να κάνει εδώ πέρα η υπηρεσία εξωτερικής δράση. Ε, ε, οι συναλφοί Δίας Δεμέρο και η Κονσουέγκρα έχουν συντάξει αυτή την έκθεση. μια ισπανική ομάδα και ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόοδος. Βλέπουμε πως με την καταπολέμηση των αιτιών γίνονται κάποια πράγματα και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να συνδέσουμε ακριβώς ε, την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα μετανάστευσης. και έτσι βεβαίω θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια λογική αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων. Δεν είναι μόνο θέμα εσωτερικής ε, πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό το είδαμε και στην ομιλία του Jean-Claude Λίντα, λοιπόν, σου παραδείω την Πρόεδρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθυστερούμε, έχουμε καθυστερήσει λίγο συναδελφοί. Είχε περικοπεί η συζήτηση αυτή σε προηγούμενη συνεδρίαση λόγω του βραβείου Ζαχάροφ. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο θέμα μας, γιατί έχουμε τις 500 τροπολογίες. Κύριε Κύριε Βαλενσιάνο, Δίας Δεμέρα, έχετε τίποτα να πείτε. Νομίζω το νόημα είναι να μιλήσουν όσοι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, Βαλενσιάνο και μετά Δίας Δεμέρα. Μόνο δύο δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα για να πω στον Πρόεδρο Μπροκ. ότι το μεγάλο συνασπισμό πρέπει να το φτιάξουμε μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο γιατί οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πολλές φορές τις αγνοούν αυτό το κοινοβούλιο. Επομένως η έκθεσή μας αυτή θα πρέπει να βοηθήσει το κοινοβούλιο να αποκτήσει και πάλι το ρόλο που πρέπει να έχει στον έλεγχο την παρακολούθηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας το Κοινοβούλιο να μιλάει με μια στεντόρια φωνή και να λέει αυτό το οποίο πιστεύουμε. Γιατί τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο τελευταίος προμαχώνας όπου γίνονται αναγνωριστεί οι, οι αναγνωριστές οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έννοια της αλληλεγγύης που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Όπως έλεγε και η κυρία Μακάβανη, η πρόεδρος. Έχουμε 550 τροπολογίες εδώ αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί στους συναδέλφους βουλευτές. Έχουμε συμφωνήσει 30 τροπολογίες ε, από τη δική μας πλευρά και έχω συμφωνήσει και με τον ε, ε, κύριο Γκερέρο από την ΤΕΒΕ να καταθέσουμε κάποιες ακόμα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με το μήνυμα που θέλει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διορθώσει από τη μια μεριά την μονομανία που φαίνεται να υπάρχει για μια αντιμετώπιση όπου υπερέχει πάντα η ασφάλεια, ο έλεγχος, η επανεισδοχή των προσφύγων, η επαναφορά τους και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεργασία κτλ. Επομένως θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η άποψη η οποία δεν βοηθάει την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει πολύ περισσότερο στον έλεγχο των συνόρων, το να μην μπορούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να έρχονται στις χώρες μας κτλ. Αυτό λοιπόν <clears throat> είναι το θέμα μια ομάδα τροπολογιών και το άλλο έχει να κάνει με την καταγγελία που εγώ θέλω να κάνω και που κάνουν και πολλοί συνάδελφοι ότι το Κοινοβούλιο όμως αυτή τη στιγμή μέσα στις δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς είμαστε στην άκρη απολύτως, ούτε καν πληροφορούμαστε όλα αυτά που γίνονται με, για το διάλογο με τρίτες χώρες. Εντάξει, είναι πολύ θετικά αυτά, αλλά θα πρέπει και εμείς να ξέρουμε κάτι. Δεν έχουμε ιδέα μέχρι που φτάνουν αυτές οι συνεννοήσεις, δεν ξέρουμε τι περιέχουν αυτές οι συμφωνίες που δίνουν την προτεραιότητα αυτό το οποίο βλέπουμε να δίνουν προτεραιότητα, σε αυτό που βλέπουμε να δίνουν προτεραιότητα είναι η επανεισδοχή των προσφύγων και ο έλεγχος των συνόρων μας. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή Ανάπτυξης και η Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων να συμφωνήσουν για το ποια θα πρέπει να είναι η φύση και ο ρόλος αυτών των συμφωνιών που τώρα υπογράφονται και που πάρα πολλές φορές γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους με τρόπο ιδιαίτερα επιδερμικό και μόνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να στείλει αυτό το μήνυμα ότι θέλουμε εμείς να ανακτήσουμε την υπεράσπιση των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι σε κίνδυνο και δεύτερον θα πρέπει να ανακτήσουμε και το θεσμικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που θέλω να προσθέσω στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Διάννη Δεμέρα Γαρσιά Συμπεθέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να δώσω μια νέα αντιμετώπιση, μια νέα οπτική γωνία, αν θέλετε, για αυτή την κοινή έκθεση. Πιστεύω ότι η ουσία της ε, εργασίας μας ήδη είχε φανεί <clears throat> στην ε, προηγούμενη αυτή συνάντησή μας που είχε να κάνει και με το βραβείο Σαχάροφ ο στόχος μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να είμαστε μετριοπαθείς μεν, αλλά συγχρόνως και φιλόδοξοι στην εργασία μας. Και να μπορέσουμε να δώσουμε έκφραση στο έργο πολλών συναδέλφων. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Βαλενθιάνο για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το τονίζουμε στην παράγραφο 19 της ε, έκθεσής μας. πρέπει να υπογραμμίσουμε και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη σημασία σε ποιοτικό και ποσοτικό που έχουν οι μαζικές μετακινήσεις των πληθυσμών, που αναφέρονται ως απλώς, απλώς ως κινητικότητα. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι μια από τις προμετωπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μαζικές μετακινήσεις, να κατανοήσουμε τις αιτίες τους, να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και την ε, παγκόσμια κοινότητα στην διαχείριση αυτών των ροών και φυσικά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προσπαθούμε να τονίσουμε τρία κριτήρια για τη διαχείριση. Ασφάλεια και τάξη, και κανονικότητα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια διαχείριση των κονδυλίων για την μετανάστευση που θα γίνεται με ένα τακτικό τρόπο. Και τονίζω το θέμα των κονδυλίων για την ε, μετανάστευση. Δεν αρκεί να έχουμε μια πολιτική ρητορική, πρέπει να έχουμε και ένα αντίκρισμα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε λεπτομέρειες στα θέματα αυτά, αλλά η δική μου προσπάθεια αυτές τις μέρες ήταν να συνενώσω κάποιες από τις τροπολογίες. Από τις 547-90 προέρχονται από το ΕΛΚ, 97 είναι από τους σοσιαλιστές, 60 από την ΑΛΤΕ, 120 από το ECR, 40 από τους πράσινους, 49 από την ΚΟΕ, 35 από την EFTD, 46 από το ENF και έχουμε διάφορες θεματικές ενότητες. Προσπαθήσαμε να τις συγκεντρώσουμε τις τροπολογίες ώστε να αλληλοενισχύονται και να μην αλληλοανερούνται. Πέραν ορισμένων λοιπόν λεπτομεριών νομίζω ότι μπορέσαμε να καταφέρουμε να έχουμε τροπολογίες συμβασμού. Θα σας αναφέρω τα βασικά θέματα, τα, τις βασικές ενότητες, γιατί είναι και η ουσία του έργου μας. Περισσότερη προστασία στις γυναίκες, στα παιδιά τα οποία είναι συνόδευτα και στη μέλη της ομάδας των ΛΟΑΔ. Ε, επίσης, περισσότερες πολιτικές μακροχρόνιου χαρακτήρα και όχι βραχυχρόνιου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο και να ανατάμουμε τις βαθιές αιτίες αυτής της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών. Πρέπει να υπάρξει αναζήτηση συγκεκριμένων και συντονισμένων δράσεων. Πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Αυτές είναι οι, οι ενότητες των τροπολογιών. Εδώ δεν θα μπω σε νομικές κατηγορίες γιατί υπάρχουν τροπολογίες που ζητούν μια διάκριση μεταξύ του τι είναι ένας πρόσφυγας ή τι είναι ένας μετανάστες και εδώ όμως δεν ξέρω αν υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αγώνας κατά της και της εκμετάλλευσης ανθρωπίνων όντων. Επίσης η δυνατότητα να υπάρξουν ασφαλείς και νόμιμες προσβάσεις, μορφές πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ είναι και το πιο αμφίμαχο σημείο που έχει να κάνει για, το, για τα υπέρ και τα κατά της συμφωνίας αυτής με την Τουρκία. Υπάρχουν επίσης τροπολογίες για την ε, ανάγκη να αλλάξουμε την αρνητική εικόνα που συνοδεύει αυτές τις ε, μαζικές μεταναστεύσεις και ακίνηση. Ε, υπάρχουν επίσης τροπολογίες για την διάλυση της λεγόμενης ζούγκλας του Καλέ. Επίσης η μεταρρύθμιση της ε, Σύμβασης του Δουβλίνου, καλύτερη συνεργασία με τις ΜΚΟ, αντιμετώπιση των συγκρούσεων και ειρήνευση μετά από αυτά, ανθρωπιστικές ε, βίζες, ανθρωπιστική διάδρομη. Όλα αυτά είναι λοιπόν θέματα τα οποία πρέπει να τα διεξέλθουμε για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα συλλέξει την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εφτά συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα διαβάσω τα ονόματα γιατί πρέπει να συντομεύουμε. Το, εκεί πέρα δεν ξέρω ποιος είναι. And then I'll tell you who, who I have... Θα σας πω ποιους έχω. Anna Gomez, um, Waldmans, Weirinen, Hautala, Corau and Epitideus. They're the names I have already. Is anybody wanting who is not the two people there, yeah, Mr. Juan Fernando, and, yeah, yeah, so it's three more. Okay. Okay, colleagues, I'm going to have to ask you for one and a half minutes maximum. Λοιπόν, 1,5 λεπτό το πολύ σας παρακαλώ γιατί έχουμε 10 ομιλητές, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να μιλήσει. Την προηγούμενη φορά δεν μιλήσαν γιατί είχαμε καθυστερήσει ούτως ή άλλως. Νομίζω πως αυτοί είναι όλοι. Και τον κύριο Λουκίε Κυρία Γκαμπριέλ. Πρώτη. Πού είναι. λοιπόν. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ για αυτό το σχέδιο έκθεση. Πρόκειται για ένα αρχικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική βάση για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι στην έκθεση αυτή δίνονται πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία. Πρώτον, παράγραφος 2, όπου προτείνεται ένα νέο μοντέλο και μια νέα αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Δεύτερον, χαίρομαι που στην έκθεση αυτή τονίζεται ότι όντως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευση και τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, προκειμένου να αποφύγουμε τις αναγκαστικές εκτοπίσεις. Τρίτον σημαντικό σημείο. Χαίρομαι πολύ για τη σημασία που δίνεται στο ρόλο που μπορεί να δραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο επιμέρους στοιχεία προς αυτό. Μια πιο συστηματική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, χρησιμοποίηση του σχεδίου δράσης της Βαλέτας και δεύτερον το να καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνίες με τις τρίτες χώρες προτεραιότητα στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων. Μεγαλύτερη ευελιξία επίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δραστικότητά της όσον αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει και για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να δίδει την έγκρισή του. Θα ήθελα να επιμείνω λοιπόν στα τρία αυτά σημεία και να προσθέσω τρία ακόμα τα οποία θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικά. Πρώτον, η έκθεση αυτή θα πρέπει να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις χώρες εκείνες, τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες επανεισδοχής οι οποίες δεν λειτουργούν. Θα πρέπει προς τις χώρες αυτές να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Δεύτερον, όπως το τονίζει και η έκθεση, τα σχέδια εξωτερικών επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα περιμένουμε όλοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει και οι ιδιωτικέ επενδύσει να λειτουργούν υπέρ των πληθυσμών εκείνων στι χώρε προέλευση και χώρε διαμετακόμιση, χώρε διέλευση. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε στις ομάδες στις οποίες αναφερόμαστε εδώ πέρα και τους, χώρες εκεί, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εκτοπίζονται εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους, για παράδειγμα στα νησιά εκείνα τα οποία έχουν καλυφθεί από το νερό της θάλασσας. Επίσης, ε, ας μην ξεχνάμε ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί μάλλον δεν θα μπορούσαν να πάρουν το καθεστώς του ε, πρόσφυγα. Αυτά τα σημεία ήθελα να τονίσω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να παραμείνει ευανάγνωστο και εύληπτο το κείμενο αυτό, να στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα και να έχει επίσης και νευσύνοπτο μέγεθος. Ευχαριστούμε. Θα δώσω... Α, το λόγο σε όσους δεν μίλησαν την προηγούμενη φορά, γιατί κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν. Λοιπόν, η Άννα Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι είναι κρίμα ότι αυτή η έκθεση δεν γίνεται μαζί με την ΛΥΜΠΕ, που είναι η επιτροπή που ασχολείται με τη μετανάστευση και το σύστημα ασύλου. Διατρέχουμε ναι, τον κίνδυνο να υπάρχει ε, να είμαστε εκτός πραγματικότητας, γιατί ωραία να μιλάμε για οικογενειακή επανένωση, αλλά αν δεν ξέρει κανείς ότι δεν λειτουργεί αυτό, ότι οι κυβερνήσεις μας δεν το σέβονται, διατρέχουμε τον κίνδυνο η έκθεση παρά τις ε, προσπάθειες που κάνουν οι συνάδελφοι να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα η έκθεση. Για να μην πω για το σύστημα επανεγκατάστασης που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Το μεγάλο θέμα νομίζω είναι ανοιχτές ε, νόμιμες και ασφαλείς δίωδοι, που δεν υπάρχει. Οπότε οποιοδήποτε, είτε πρόσφυγας είτε μετανάστης, ε, ε, έρχεται παρανόμως στην Ευρώπη γιατί δεν υπάρχουν ασφαλείς ε, και νόμιμες δίωδοι. Δεν το κάνει αυτό καμία χώρα. Ακόμα και αυτή η μπλε κάρτα που έχουμε υποτίθεται δεν λειτουργεί. Έχουμε και μια σχετική έκθεση στη Λίμπε. Το ερώτημά μου είναι το εξή προς τους συγητές. Μπορούμε να είμαστε έτσι συνεκτικοί και να κάνουμε κάποια διαφορά. Δηλαδή, η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάνουν διμερείς διαπραγματεύσεις αγνοώντας το Κοινοβούλιο με το σύμφωνο αυτό μετανάστευσης που παρέκαμψε τελείως το Κοινοβούλιο. Π.χ. μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι τέρος στον αντιμετωπίσει τις αιτίες ε, διοικείται από μια ελίτ ε, η οποία δημιουργεί τελικά πρόσφυγες και μετανάστες. Μιλάω για την Αιθιοπία, γιατί δεν είναι η μόνη. Ή τώρα μας λένε ότι έχουμε μια συνεννόηση με το Αφγανιστάν. Ε, και ως αν επρόκειτο μια ασφαλή χώρα όπου μπορούν να επιστραφούν οι άνθρωποι και οι περισσότεροι συνοδευτοί ανήλικοι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι Αυγανοί λόγω της τρομερής κατάστασης που επικρατεί εκεί ειδικά όσον αφορά τη μειονότητα των Χαζάρων. Όπως είπε και ο Αντώνιο Γκουτιέρες, οι μόνοι που κάνουν κάτι είναι οι διακινητές, γιατί εκμεταλλεύονται την κατάσταση και το ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις αιτίε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Λοιπόν, Γιώργο και για το ECR. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή κυρίως ε, θα πρέπει να αναφερθεί στην πολιτική ευθύνη για αυτή τη μεταναστευτική κρίση. Πρέπει να αναφερθεί αυτό. Η άνοδος της ε, παράνομης μετανάστευσης σημαίνει και αύξηση των ανθρωπίνων τραγωδιών και των προβλημάτων. Βλέπουμε όλο και περισσότερες τραγωδίες κατά την ε, διαδρομή και η ευθύνη για την κορύφωση αυτής της κρίσης οφείλεται σε κάποιες κυβερνήσεις κρατών μελών και αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν αντιλαμβάνουμε γιατί μιλάμε, ε, δεν μιλάμε για την υποχρέωση ε, καταπολέμησης ε, της ε, παράνομης μετανάστευσης. Εδώ και 1,5 χρόνο ήδη είχαμε τις πρώτες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κρίση αυτή. Και ήδη τότε το Συμβούλιο έλεγε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει υπηρεσία εξωτερικής δράσης μέσω των κρατών μελών μια έντολη για να διαχειριστεί ε, αυτό το θέμα. Τρίτον, τώρα προτείνεται μια ενιαία ε, μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα βγήσει σε ε, ακόμη περισσότερα προβλήματα. Είμαστε ήδη σε πολιτική κρίση μετά το Brexit ούτως ή άλλως. Και τελευταία παρατήρηση, όταν μιλάμε για οικογενειακή επανένωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για χώρες όπου το αστικό δίκαιο επιτρέπει την πολυγαμία. Οπότε μιλάμε για υπήκους κρατών που έχουν διαφορετικό σύστημα δικαίου. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ε, το θέμα αυτό είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ε, αντιλαμβάνομαι την κυρία Ντόμες που λέει πως ίσως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα μπορούσε εκεί να είναι κάπως πιο σοβαρή η έκθεση. Κοιτάξτε, για εμάς θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η έκθεση, να έχουμε ένα σχέδιο, να πούμε πώς φανταζόμαστε εμείς ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και έχουμε καταθέσει κάποιες σχετικές απολογίες για να γίνει συγκεκριμένη αυτή η έκθεση. Ένα από τα σημεία στα οποία έχω αναφερθεί εγώ αφορά το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων όσον αφορά την υποδοχή, αλλά να σας πω και το εξής. Η Europol λέει ότι αυτή τη στιγμή αγνοούνται 10.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι θα κάνουμε για να βρούμε αυτά τα άτομα μπορεί να πρόκειται για άτομα τα οποία δεν έχουν και τόσο αγαθές ε, προθέσεις. Επίσης ε, να αναφερθώ στην ε, ζούγκλα του Καλέ. Θα είδατε φαντάζομαι τι έγινε, πήγα και εγώ επί τόπου να δω το τι έγινε. Τι γίνεται λοιπόν, το διέλυσαν εκεί πέρα τον καταβλισμό και ξεφυτρώνουν αλλού καταβλισμό. Τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στην Αγγλία, τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Ο κόσμος περιμένει μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για το θέμα αυτό, ειδικά για τα παιδιά. Και πραγματικά αυτό το οποίο είδα στο Καλέ δεν είναι αντάξιο της ε, Ευρώπης και δεν επιτρέπεται να ξανασυμβεί αλλού. Και κάτι άλλο ακούστηκε και κάτι για τις ε, νόμιμες ε, διόδους. Πράγματι πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να ε, έχουμε μια καλή εκτίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, το χρόνο σας παρακαλώ. Η κυρία Χάουτολα. Yeah, thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει κατά προτεραιότητα να πετύχουμε είναι να έχουμε μια μετανάστευση, μεταναστευτική πολιτική που να βασίζεται στο ανθρωπιστικό δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί αυτό και στην έκθεση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πάντα στη σωστή τους διάσταση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πρόσφυγες, μάλλον οι πρόσφυγες είναι 0,2%. Ας το συγκρίνουμε αυτό με το ποσοστό προσφύγων στο Λίβανο, 20% για παράδειγμα, ή στην Ιορδανία, εξίσου σημαντικό ποσοστό. Είμαστε μια οργανωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανωμένες κοινωνίες, οργανωμένα κράτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινή ευθύνη και ένα κοινό επιμερισμό όσον αφορά την προσφυγική αυτή κρίση. Τα νέα μέσα τώρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κάποιες προποθέσεις όσον αφορά την επανεισδοχή, την, απο, την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι χρησιμοποιούμε μέτρα αναπτυξιακής συνεργασίας που προκαλούν τελικά περισσότερα προβλήματα και περισσότερα βαθύτερα αίτια, αν θέλετε, για την αύξηση της μετανάστευσης. Τέλος, χρειαζόμαστε έναν πολύ αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο και χαίρομαι που ο κ. Δίας Δεμέρα αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, διαφορετικά δεν θα υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο στον τομέα τη διαχείριση, τη μετανάστευση και τη προσφυγική κρίση. Θα έχουμε όλο και περισσότερε ανεπίσημε συμφωνίε, όπω μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφγανιστάν ή όπω έχουμε δει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει παγιωμένο δομικό μοντέλο συνεργασία με τρίτε χώρε για τη διαχείριση τη μεταναστευτική κρίση. Ανταυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει τις συμφωνίες αυτές, να ασκεί δηλαδή δημοκρατικό έλεγχο, δεν μπορεί να παρακάμπτεται ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, Μα καλέσαμε την Επιτροπή Λιμπέλη στα πλαίσια του άρθρου 55, αλλά δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είχαν πάρα πολύ φόρτο εργασία. Άρα θα γνωμοδοτήσουν. Ο κύριο Ιγνάθιο Κοράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μετά όσα είπαν οι προλήσαντες και κυρίως η προελίσσασα όσον αφορά το πολύ αυξημένο ποσοστό το οποίο έχουμε σε άλλες χώρες και το μικρό ποσοστό τελικά προσφύγων σε σχέση με τον κοινοτικό πληθυσμό εμείς ε, θα πρέπει με το μικρό αυτό ποσοστό προσφύγων να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ανταυτού, να παρουσιάσουμε τα πράγματα ως απόλυτη καταστροφή και δεν μπορούμε τελικά να συντονιστούμε. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω και με τη συνεργασία της ΛΥΜΠΕ να καταφέρουμε να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι λειτουργούν εντελώ εγωιστικά και εθνικιστικά ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι πολύ καλή για ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε που θέτουν ω προτεραιότητα κάποιε πτυχέ του ζητήματο. Για παράδειγμα, τονίσουμε περισσότερο ότι δεν υπάρχει απαραίτητη άμεση πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε τρίτες χώρε όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο. Αναφερόμαστε περισσότερο στα βαθύτερα αίτια. Δεν μπορούμε απλώ να αντιδρούμε. Πρέπει ω Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να προλαμβάνουμε τι καταστάσει αυτέ και να αποτρέπουμε τελικά τα φαινόμενα εκείνα τα οποία οδηγούν σε αυξημένε μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ροέ. Κάτι ακόμα το οποίο τονίζουμε είναι το ζήτημα της πάταξης της διαφθοράς. Γίνεται πολύ μικρή αναφορά στο κείμενο αυτό, πιστεύοντα αυτό ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το ζήτημα της πάταξης διαφθοράς προκειμένου να υπάρχουν ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης στις τρίτες χώρες και προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν εκεί. Όσον αφορά τα πρότυπα, προφανώς θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους εγωισμούς που εκφράζουν αυτή τη στιγμή ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τα όσα λέγονται για τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Είναι ένα λαθασμένο ημίμετρο, θεωρώ, το οποίο δεν λύνει πραγματικά την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ουσιαστική μετανα... Ε, συνεργασία με τις τρίτες χώρες και να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τελικά τα δίκτυα της παράνομης διακίνησης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι συνθήκες ισχύουν στις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και αν καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι εκεί θα μπορούσε να γίνει και μία αναφορά στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Εν συντομία αυτές είναι οι τροποποιήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ κύριο Επιτίδιος, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εάν θελήσουμε να εξετάσουμε την ε, έκθεση ως ένα φιλολογικό κείμενο, τότε οπωσδήποτε θα μπορούσαμε να το βαθμολογήσουμε με άριστα. Αν θέλουμε όμως να το δούμε ε, ως μια πραγματική προσπάθεια αντιμετωπίσεως του προβλήματος το οποίο έχουμε, τότε οπωσδήποτε ε, θα το χαρακτηρίσουμε ως ένα απλό ευχολόγιο. Δεν το λέω αυτό με ειρωνική διάθεση, αλλά με πραγματιστική. Βλέπετε, η αλλοπρόσαλη πολιτική που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, από μια μεριά πολιτική ανοιχτών συνόρων και τώρα ε, έλεγχος συνόρων, ε, πανικός γενικός διότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ε, ροή των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι εξέλεγκτη. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη ροή των μεταναστών όταν δεν, ε, δεν συνεργαζόμαστε με τα κράτη τα οποία είναι οι χορηγοί, είναι οι πηγές της ε, ροής των προσφύγων. Η κυρία Γκόμες ανέφερε την Αιθιοπία, εγώ δεν θα κομίσω γλάφκα εις Αθήνα σαν σας αναφέρω την Τουρκία και όλα αυτά ε, ε, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Βλέπετε οι ορισμένες χιλιάδες μεταναστών, παρανόμων μεταναστών δημιούργησαν τη ζούγκλα του Καλέ. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot. Γνωρίζετε γιατί πολλέ και πολλοί από εσά έχουν επισκεφτεί τα hot spot στην Ελλάδα, ποια κατάσταση επικρατεί εκεί. Ε, συγκλοκές μεταξύ διαφόρων, μεταναστών διαφόρων εθνών, βιασμοί γυναικών, ε, παιδιά τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, απροστάτευτα και όλα αυτά θέλουμε εμείς να τα ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εάν προηγουμένως δεν αποφασίσουμε να μοιράσουμε, να σταματήσουμε καταρχάς τη ροή των προσφύγων προς τις ε, ε, χώρες της Ευρώπης και παράλληλα την κατανομή των ήδη υπαρχόντων με την αναλογία η οποία μπορεί να αποδοθεί σε κάθε κράτος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, όπως είναι σαφές. Είμαστε πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον την ε, κοινή αυτή ενέργεια της ε, Επιτροπής ε, Ανάπτυξη, ε, και εξωτερικών υποθέσεων, αλλά εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε και το θέμα αυτό και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ των Δημοσίων Ελευθεριών. Εγώ θα ήθελα να σκεφτώ περισσότερο για τη διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο μια Επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει στις ε, εκθέσεις μιας άλλης Επιτροπής. Η κυρία Βαλεντιάνο τόνισε ότι το ουσιαστικό είναι να έχουμε μια κριτική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου που αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την πίεση λεγόμενης μεταναστευτικής κρίσης και είναι μια πολύ αρνητική στροφή αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι είπε σε σχέση με τη συμφωνία με την ε, Τουρκία. Ο κ. Δίας Δεμέρα μίλησε για τη δήλωση σε σχέση με την Τουρκία, γιατί ακούσαμε θετικές δηλώσεις από την Κομισιόν ότι λέει ότι αυτή η συμφωνία καταφέρνει να μειώσει τις ροές προσφύγων από την ε, <clears throat> Τουρκία, αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι έχει μεταφέρει το θέμα στις βορειοαφρικανικές ακτές, στην άλλη όχθη της Μεσογείου, όπου χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συσσωρευτεί γιατί έχει μεταφερθεί εκεί το πρόβλημα. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, είναι αυτό που είπε πάλι και ο κύριο Δίας Δεμέρα, που είναι το, η σημασία που έχουν οι λεγόμενοι ασφαλείς και νόμιμοι διάβροι Να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για νόμιμη μετανάστευση, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή απλώς που κάνουμε αυξάνει την απόγνωση αυτών των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, που δοκιμάζουν την ζωή τους για να μπορέσουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και μετά έχουμε και τον κώδικα της βίζας. Όλα τα ψηφίσματα λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στην πολιτική μας. Εμείς έχουμε πει πως είμαστε υπέρ μιας ανθρωπιστικής βίζας, αλλά τον μπλοκάρει συνεχώς το Συμβούλιο, μη λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε υπέρ ε, της ε, ανθρωπιστικής ε, βίζας. Κύριε Λούκε, σας παρακαλώ να είστε πολύ ε, σύντομος γιατί μιλήσατε και στην προηγούμενη Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Να αφαιρθώ σύντομα σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάουταλα, γιατί είναι χαρακτηριστικά του ότι σε αυτή την έκθεση Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι περισσότερο στον, στη σφαίρα των ιδεωδών και μακριά από τον ρεαλισμό. Μιλάτε για ένα 0,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να δούμε πως υπάρχει μια ανισοκατανομή. Στη χώρα μου 20% του πληθυσμού έχει μια καταγωγή μεταναστευτική. Ε, οπότε υπάρχουν περιοχές ε, στις οποίες ε, είναι 30 ή 40% του πληθυσμού. Και με δεδομένα τέτοια νούμερα δεν μπορούμε να λέμε έτσι απλά πόσο επιθυμητή είναι η περαιτέρω μετανάστευση, αλλά να δούμε τα πραγματικά προβλήματα. Ειδικά όταν μιλάμε για άτομα από την Τουρκία ή από τις αραβικές χώρες γνωρίζουμε ότι έχουν δυσκολίες να ενταχθούν και 20-30% αυτών δεν έχουν ε, κάποια, δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση και βεβαίως αυτό σημαίνει πως μετά αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα. και καλωσορίζω αυτό το οποίο υπόθηκε πως ε, θα πρέπει πράγματι η έκθεση να αντικατοπτρίζει την άποψη των βουλευτών. Σας ευχαριστώ και Ζωάννη που δεν μίλησε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το θέμα αυτής της έκθεσης είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και της προσβυγικής κρίσης. Εγώ είμαι σκιώδης της από την Άλτε στην Επιτροπή Άλτε και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική πολιτική είναι σωστή αυτή η, η πρόταση, αλλά υπάρχει και η πτυχή των εξωτερικών θεμάτων. Εγώ έχω κάνει δύο τροπολογίες που λέω ότι καταρχήν ότι οι στρατιωτικές κρίσεις και η βία είναι η κύρια αιτία αυτής της κρίσης μετανάστευση και προσφύγων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει την ΑΦΕΤ η οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει ειρηνική επίλυση αυτών των συγκρούσεων. Και η δεύτερη πρότασή μου τροπολογίας έχει να κάνει με την ιδέα ότι έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τους φορείς του ΟΗΕ και με τις γειτονικέ χώρες, να φτιάξουμε κέντρα υποδοχής και κέντρα υποδοχής προσφύγων υψηλού επίπεδου, όπου προσπαθούμε να δώσουμε στα άτομα αυτά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το δικαίωμα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άτομα αυτά μετά θα πρέπει να έχουν αυτό το δικαίωμα. Έτσι θα μπορέσουμε, αν έχουν το δικαίωμα, θα έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα σταματήσουμε την ε, αλόγιστη και ανεξέλεγκτη ροή και τους θανάτους που βλέπουμε στην ε, Μεσόγειο. Νομίζω ότι αυτές οι δύο τροπολογίες <clears throat> πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι στην αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής ΑΦΕΤ που ενδιαφέρει για αυτή την έκθεση. Ο Γκερέρο Σαλόμ, για ένα λεπτό μοναχανέ, ναι, ευχαριστώ πολύ. μετά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Λόπες, νομίζω ότι είναι σαφές ότι χρειάζεται μια αλλαγή στη, στο αφήγημα, όχι αλλαγή μόναχα σε στάση, κατά των προσφύγων, αλλά και για τον τρόπο που βλέπουμε τους πρόσφυγες. Υπάρχουν μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά για διαφορετικούς τρόπους. Η μετανάστευση είναι μια τάση του καιρού μα, αλλά οι πρόσφυγες είναι απόρρια των συγκρούσεων. Θα πρέπει εμείς να εμποδίσουμε τις συγκρούσεις αυτές με μια σωστή αντιμετώπιση στον εξωτερικό τομέα ω ένα παγκόσμιο παίκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαι ο μόνιμος εισηγητής για τα θέματα ανθρωπιστική δράση, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο <clears throat> δεν είναι μονάχα θέμα. Νοοτροπία είναι ένα θέμα πραγματικότητα και εξάλλου δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την έκθεση αυτή λέγοντα ότι ένα πράγμα λέει η έκθεση και κάτι άλλο λέει η πραγματικότητα. Γιατί αυτό το οποίο θέλει η έκθεση να κάνει ακριβώ είναι να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα που έχουμε ενώπιον μα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών. Έχω μονάχα δύο παρατηρήσει να κάνω η ίδια. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω τις ανησυχίες των συναδέλφων που, που γίνεται χρησιμοποίηση αναπτυξιακών κονδυλίων για μία βραχυπρόθεσμη και μόνο αντιμετώπιση κρίσεων όπως είναι η τρέχουσα κρίση. Είδαμε χρήματα για την ε, ε πρόθεση της δημοκρατίας και άλλα τέτοια να μεταλαμπαδεύονται για την αντιμετώπιση της κρίσης και επίση με τι συμφωνίε που γίνονται για τη μετανάστευση δίνουμε σε άλλες χώρες μοχλου πίεση εναντί τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή παραγωγικά να επικρίνουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία <clears throat> γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μοχλούς πίεση απάνω μα σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική, τον έλεγχο μεταναστευτικών ροών. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν <clears throat> και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα σας παρακαλέσω να είσαστε <clears throat> σύντομοι. Δίνω το λόγο στον ε, Διευθυντή της Διζιντεύκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μας δείτε τη δυνατότητα να πάρουμε το λόγο στη συζήτηση αυτή. Συζήτηση πάρα πολύ σημαντική και πολύπλοκη όμως αρκεί να ακούσουμε του ευρωβουλευτέ που πήραν το λόγο και συνειδητοποιούμε πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα. Μιλάμε για συγκρούσει, για κρίσει. Αναφερόμαστε σε λόγου για του οποίου ορισμένοι θέλουν να εγκαταλείψουν τι χώρε που να έρθουν στην Ευρώπη. Ας είμαστε λοιπόν πολύ, πολύ προσεκτικοί. Α μην μπερδεύουμε όλους αυτούς διαφορετικού λόγου. Θα έκανα λοιπόν καταρχά μία έκκληση. Αν πραγματικά θέλετε να κάνουμε μία αξιοπρεπή συζήτηση του ζήτηματο, τότε θα πρέπει να βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε παρκώ το ζήτημα αυτό. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση μέσα σε μισή μόνο ώρα να κάνουμε πλήρη συζήτηση και να, τα, να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Εμείς σαφώ θέλουμε να σα δώσουμε περισσότερε πληροφορίες, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρακάμψουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώ διατηρεί σε πάρα πολλού τομεί ε, το δικαίωμα ελέγχου, δημοκρατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου τονίστηκε αυτό και από κάποιους ομιλητές, αυτό προβλέπεται σε κάποιους τομείς από συγκεκριμένη νομική βάση, σε άλλους πάλι τομείς δεν προβλέπεται ακόμα. Θα μπορούσαμε πάντως ε, εμείς να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά να πρόκειται σε εσά να καλείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να μπορούμε να συζητούμε με εσά τα ζητήματα αυτά επαρκώς. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο στην παρέμβασή μου ετέθηνε ερώτημα εταιρικών σχέσεων και εταιρικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Αυτό αποφασίστηκε στη Σύνοδο της Βαλέτα, ότι δηλαδή σε σχέση με τις χώρες της Αφρικής, για παράδειγμα, θα έχουμε μια κοινή προσέγγιση στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για εταιρική σχέση, ουσιαστική εταιρική σχέση. Και όντως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα θετικό αφήγημα, το είπατε πολύ, Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και από τη θετική του μόνο πτυχή. Να έχουμε ένα θετικό αφήγημα, να βλέπουμε ποια είναι η προσφορά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες αυτές, προκειμένου να διαχειριστούν οι χώρες αυτές καλύτερα τη μετανάστευση. Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι να σταματήσει αναγκαστικά η μετανάστευση, αλλά να την χάνει καλύτερης διαχείρισης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρηματοδοτούμε τις χώρες αυτές για να αντιμετωπίσουμε και τα δεινά των χωρών αυτών. Κακή διαχείριση, δεινή οικονομική, δια... Ε, δεινή οικονομική κατάσταση και το καθεξής. Θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο για την Αφρική, το καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, που αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Σε καμία πρόθεση, σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από την πολιτική ανάπτυξη για ζητήματα που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Ξέρετε όμως ότι η μετανάστευση αναγνωριζόταν ανέκαθεν και εξακολουθεί και αναγνωρίζεται όσα κριτήριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν η μετανάστευση να αντιμετωπιστεί θετικά, να την εκμεταλλευτούμε εντό εισαγωγικών θετικά αν θέλετε, προκειμένου μέσω της μετανάστευσης να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και σε πολιτικό επίπεδο. Το τελευταίο διάστημα, επίτροποι, υπουργοί, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν πάει σε ορισμένε τρίτε χώρε προκειμένου να θεσπίσουν εκεί μια εταιρική σχέση, έναν διάλογο, ο οποίο δεν υφίστατο στο παρελθόν. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο και να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, ακόμα και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει και για τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχουμε αρχίσει να δεσμευόμαστε με χώρες όπως η Τουρκία αλλά και με άλλες χώρες σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν αναφέρεται σε αυτό βέβαια η έκθεση είναι το τι γίνεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό ασχολούνται οι συνάδελφοι οι αρμόδιοι για την εσωτερική πολιτική. Και από αυτού όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολλοπλοκότητα του ζητήματος. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε επιμέρους τμήματα του ζητήματος αυτού ή να επιμερίσουμε αρμοδιότητες από τη μία επιτροπή στην άλλη. Εμείς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερική δράση, προκειμένου να καταφέρουμε να δούμε το πρόβλημα σφαιρικά, τα στοιχεία από την εξωτερική πολιτική, την εμπορική πολιτική, την επενδυτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια ολιστική σφαιρική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματο. Και αυτή είναι η μόνη επιλογή τελικά. Δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε, δεν μπορούμε προφανώ να κλείνουμε τα σύνορα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών έχει υποβάλει πάρα πολλέ προτάσει. Πολλέ φορέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη δυνατούν να ακολουθήσουν τον έντονο αυτορυθμό ρυθμό ανάληψη πρωτοβουλειών από τα δύο αυτά όργανα. Το λέω όμω αυτό για να σα πω ότι προσπαθούμε να δρούμε προδραστικά. Προσπαθούμε να προλάβουμε την ε, εμφάνιση περαιτέρω αρνητικών καταστάσεων και προσπαθούμε να συνδυάσουμε την μεταναστευτική πολιτική με τις υπόλοιπες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χειριστούμε καλύτερα την κατάσταση. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που εξέθεσαν οι ευρωβουλευτές. Πρέπει σαφώς να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Θα έχουμε του χρόνου, του 2017, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μία σύνοδο με τις χώρες της Αφρικής. Ας την προτιμάσουμε καλά τη σύνοδο αυτή. Ας στηρίσουμε μία επικοδομητική στάση. Πιστεύω ότι το μεσανατολικό κάποια στιγμή θα επιληθεί, αλλά το ζήτημα της μετατόπισης πληθυσμών και της αύξησης του πληθυσμού της Αφρικής δεν πρόκειται μία νυχτή να επιληθεί. Πρέπει λοιπόν ήδη από τώρα να αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις ε, του μέλλοντος. Για όλα αυτά θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίρια Μπρούσκα Πίνο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τώρα έχει το λόγο. Good evening. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια μόλις έκανε ο κ. Ρουδιχάζερ και να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία που είναι σημαντικά στη συζήτηση αυτή του του λεχθέντος και καθώς η έκθεσή σας αναφέρει κάποια πράγματα η μετανάστευση είναι πλέον γεγονός και θα πρέπει να την διαχειριστούμε είναι σαφές πως ανεξαρτήτως των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, σαφώς ε, απαιτείται μια μακροπρόθεσμη αντίδραση η οποία θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στην πολιτική της Ένωσης και όπως ε, υπόθηκε για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο εταιρικών σχέσεων που ξεκίνησε φέτος με πέντε χώρες προτεραιότητας στην ε, υποσαχάρια Αφρική. Οπότε έχει ενσωματωθεί ε, στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων που θέλουμε να αναπτύξουμε και αναπτύσσουμε με τις χώρες αυτές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι καινούρια θα έλεγα το ένα είναι η μέθοδος ε, εργασίας, ο συντονισμός μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών και όπως είπε και ο Ρίτι Χάζερ πρόκειται για έναν διάλογο άνευ προηγουμένου με τις πέντε χώρες προτεραιότητας όπου και τα θεσμικά όργανα, οι επίτροποι, η υπατή εκπρόσωπος και οι αρχές των κρατών μελών έχουν επαφές με τις ε, χώρες ε, εταίρους για να συζητήσουμε ζητήματα μετανάστευσης στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής δεύτερον. Η προσέγγιση δεν είναι, όπως είπαμε, μόνο βράχη πρόθεσμη. Γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις και είναι συνολική και ολιστική θα λέγαμε η παγκόσμια προσέγγιση λοιπόν για τη μετανάστευση και την κινητικότητα που αντιμετωπίζει το θέμα <coughs> της νόμιμης μετανάστευσης και κινητικότητας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ζητήματα ασύλου και ζητήματα ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως είπα μπαίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τρίτον, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει η πολιτική εμπλοκή και όπως θα δείτε και στην έκθεση πρόοδου που δημοσίευσαμε τον προηγούμενο μήνα η προσέγγιση αυτή ε, αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον από τις χώρες εταίρους και βλέπουμε κάποια ανταπόκριση. Τέλος θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για να ξεκαθαρίσω πως τα σύμφωνα αυτά δεν είναι συμφωνίες, ε, είναι μια διαδικασία αμοιβαίας πολιτικής ε, επαφής με τις χώρες αυτές ε, με στόχο να δημιουργηθεί ένας ενάρετος, θα έλεγα, κύκλος. Και όπως είπα το θέμα πηγαίνει πέρα από τις επιστροφές ε, και τους επαναπατρισμούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν θα προκύψει τίποτα αν μείνουμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να υπάρξει, όπως είπα, μια συνολική αντιμετώπιση. Και τέλος, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Η συνέχεια που θα δοθεί στις ε, συνόδους κορυφής του Σεπτεμβρίου υπάρχει τώρα μια δήλωση της Νέας Υόρκης για τους ε, πρόσφυγες και μετανάστες ε, την οποία συνυπέγραψαν 193 χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού και θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις τώρα που έχουμε αναλάβει με τις χώρες εταίρους και είναι νομίζω μια σημαντική αφετηρία για να υπάρξει, όπως είπα, μια παγκόσμια συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα σε τρεις εβδομάδες. Οι συνεισηγητές έχουν να πούν κάτι τώρα ή μπορούν να περιμένει. Κύριε Δίας, δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα όλες τις ε, παρεμβάσεις που έγιναν και από την Κομισιόν και την Εξωτερική Υπηρεσία και από τους συναδέλφους για την συμμετοχή της ΛΥΜΠΕ. Η ΛΥΜΠΕ συμμετέχει σε αυτή την έκθεση. Η κυρία Βερζιά θα δώσει τη γνωμοδότηση από την πλευρά της ΛΥΜΠΕ σε αυτή την έκθεση. Και δεύτερον, αναφέρομαι σε αυτά που είπε η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας εξωτερικών, εξωτερικής δράσεως. Και είναι, είπε ότι είναι ανοιχτή στην συμβολή του Κοινοβουλίου και υπάρχει και νομική βάση για όλα αυτά. Το λέμε και στην εκθέσή μας. Υπάρχει μια νομική βάση και αυτό είναι σημαντικό για την εκθέση αυτή, το οποίο μας καλύπτει εμάς η συνθήκη για τη λειτουργία ε, λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης τα άρθρα 218 και 216. Αλλά επίσης θα πρέπει να θυμηθούμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών για την ε, μετανάστευση και του Συμβουλίου Ανάπτυξης, αλλά επίσης και ένα σύνολο εκθέσεων από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολογισμών και της Επιτροπής ε, ε Ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν <clears throat> είναι η βάση του έργου μας, αλλά όλα αυτά σημαίνουν ότι εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε όχι μόνο ένα ρόλο του Κοινοβουλίου με τρόπο απόλυτα τεκμηριωμένο και δικαιολογημένο, αλλά να τονίσω ότι έχουμε νομική βάση απολύτω για αυτό το λόγο. Η, κυρία Βαλεντιάνο. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία είπε ο κύριε Στιάς Μέρα έχουμε νομική βάση, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι συμφωνίες μπορεί να μας αφήνει στην άκρη, αλλά γίνονται κάποιες ενέργειες στις οποίες δεν τις συμμετέχει, δεν τις συμμερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι με το να εκφράσουμε την άποψή μας με ένα διάφορο τρόπο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει καταρχήν να αποφύγουμε να έρχονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ευρώπη και αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο καλύτερος τρόπος να το κάνει είναι με το να συνεργαστεί με κάποιες από τις χώρες <clears throat> και με κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν έχουν εχέγγυα για τον ελάχιστο σεβασμό στα ανθρωπίνα δικαιώματα. Αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα γιατί εμείς συνεργαζόμαστε με χώρες οι οποίες από άλλες απόψεις έχουν επικριθεί ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα πρόβλημα συνέπεια το οποίο είναι ουσιαστικό. Λέμε ότι θέλουμε να αποφύγουμε να έρχονται οι πρόσφυγες από την αρχή, αλλά ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό εμποδίσουμε ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να πάνε να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα λέμε ότι όταν υπάρχει πόλεμος δεν είναι μετανάστες, όταν υπάρχει κλιματική αλλαγή δεν είναι πρόσφυγες κτλ. Όχι. Εμείς όμως έχουμε κανόνες του δικαίου και αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το Κοινοβούλιο φοβάται ότι αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Φοβάμαι ότι γίνονται συμφωνίες επονίδιστες με κυβερνήσεις με τις οποίες εμείς δεν θα έπρεπε να κάνουμε τέτοια συμφωνία στο αν υπάρχει νομική βάση ή όχι, δεν έχει σημασία. Θα το δούμε. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Είναι πολλοί οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμφωνούν με αυτά που κάνουμε. Όπω παραδείγματο στην περίπτωση συμφωνία με το Αφγανιστάν, που είναι όνειδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο αυτή. Ξέρω ότι είναι πολύπλοκο το πρόβλημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Αλλά προσέξτε γιατί παίρνουμε αποφάσει οι οποίε σε πάρα πολλέ περιπτώσει απέχουν πολύ από τις υποχρέωσεις που έχουμε εμείς ως βουλευτές που είναι να σεβαστούμε και να είμαστε υπέρμαχοι των αξιών χάρη στις οποίες υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να συμμετάσχει με πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο διάφορο τρόπο και αν μπορέσουμε να εμποδίσουμε κάποιες από τις ολιστήσεις που γίνονται από την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ίσως όχι, αλλά κυρίως από το Συμβούλιο, ας το κάνουμε γιατί αυτό είναι πράγματι είναι υποχρέωσή μας δίνω στο συμπρόεδρο μου για να κλείσει το λόγο. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση, η οποία θα είναι πολύ χρήσιμη για τους ε, συνεισηγητές μας. Η επόμενη κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών θα είναι 28-29 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε και τους διερμήνες που έδειξαν μεγάλη ευελιξία.